Przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καθίστε σας παρακαλώ. Ah, Otwieram posiedzenie. Κυρίσω την έναρξη της Συνόδου. Επαναλαμβάνεται η σύνοδος ομιλίας που διακόπη τη 7η Απριλίου 2010. Καθίστε σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Proszę και κύριοι, έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης της 7 Απριλίου 2010. Έχετε παρατηρήσει από αυτόν, όχι. Θεωρούνται λοιπόν τα πρακτικά εγκεκριμένα.